λαμβάνονται και στα προγράμματα του Z20 και Z8. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψήφιση επίσης και της πρότασης ψηφίσματος που έχει κατατεθεί από την πρόεδρο Ζολή όπως είπα θα ψηφιστούν αύριο το μεσημέρι 12.00 και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη που σίγουρα θα είναι το πρώτο που θα έχει έναν άνδρα εισηγητή στην απόψινή μας συνεδρίαση που είναι του κυρίου Παπαστάμκου αυτή η έκθεση και είναι η γεωργία το θέμα και το διεθνές εμπόριο. Θα λάβει τον λόγο εισηγητής. Τέσσερα λεπτά κύριε Παπαστάμκο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ένωση εξετάζει το μέλλον της ΚΑΠ, η εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου καθίσατε έτσι περαιτέρω ουσιώδης. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας ζητείται να συνεισφέρει ένα και περισσότερο στην παραγωγή δημοσίων αγαθών μέσω αυστηρών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και ευζοίας των ζώων animal welfare. Είναι λογικό λοιπόν ότι οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων οφείλουν να παρέχουν τις ίδιες εγγύησεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον ποε η ένωση τηρεί επιμακρών και ως ένα βαθμό εξακολουθεί να τηρεί αμυντική στάση όσον αφορά τη γεωργία. ωστόσο θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τη ριζική αναθεώρηση της καπ. η ένωση έχει μειώσει δραστικά σε αντίθεση με άλλους σημαντικούς εταίρους τις ενισχύσεις που οδηγούν σε στρέβλωση του εμπορίου. Έχει επίσης προβεί μονομερός σε δραστική μείωση των εξαγωγικών επιστροφών ενώ ανταγωνιστικοί εμπορικοί εταίροι εξακολουθούν να κάνουν εκτεταμένη χρήση άλλων μορφών εξαγωγικών κινήτρων. Ακόμη η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. η ένωση έχει ήδη προβεί σε μια εξαιρετικά γενναιόδορη προσφορά offer στις γεωργικές διαπραγματεύσεις η οποία ωστόσο δεν ανταποδόθηκε μέχρι σήμερα με ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας από άλλες ανεπτυγμένες και προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. ταυτοχρόνως η κομισιόν διεξάγει διμερείς και διαπεριφερειακές διαπραγματεύσεις με πολυάριθμους εμπορικούς εταίρους. Ο αντίκτυπος στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα όλων των επιμέρους γεωργικών παραχωρήσεων παράλληλα με τις εκκρεμείς γεωργικές διαπραγματεύσεις μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Στο πλαίσιο αυτό, κυρία Επίτροπε, καλούμε την Κομισιόν να διαφυλάξει τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας της ένωσης καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο ε, γεωργικών προϊόντων διατροφής το οποίο αποτελεί στρατηγική συνιστόσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. επισημαίνουμε ότι οι παραχωρήσεις εις βάρος της γεωργίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελούν το αντάλλαγμα monnaie change, έναντι της αυξημένης πρόσβασης στις αγορές βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουμε την ανάγκη μελέτης αντικτύπου η οποία να προηγείται της έναρξης διαπραγματεύσεων και σε κάθε περίπτωση της ανταλλαγής προσφορών. η κομισιόν καλείται επίσης να προωθήσει τα επιθετικά συμφέροντα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτουν τα υψηλής ποιότητας γεωργικά είδη διατροφής της ένωσης. ιδίως δε να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων εκ μέρους των εταίρων μας τόσο στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών συμφωνιών όσο και στο πλαίσιο της ακτα και του ποε. συμπερασματικά η γεωργία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζωνος σημασίας για το κοινωνικό σύνολο ο φεδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω των αγορών. συνεπώς η κύρια πρόκληση συνίσταται στον αποτελεσματικό συνδυασμό εμπορικών και μη εμπορικών παραμέτρων. ως εκ τούτου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η οικονομική γεωγραφία της καπ καθιστά επιτακτική την ανάγκη αυξημένης συνοχής μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου της ένωσης μεταξύ γεωργικής πολιτικής εσωτερικών πτυχών της κοινή αγροτικής πολιτικής και των εξωτερικών πτυχών ή αν θέλετε μεταξύ του αυτού που λέμε in foro interno και in foro externo δηλαδή της παρουσίας της ένωσης στην παγκόσμια εμπορική κλίμακα στις δύο εκφάνσεις της την διμερή και την πολυμερή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Δραχθήκατε της ευκαιρίας ε, ότι πραγματικά το χρονόμετρο ήταν, ξέφυγε κάπως, ήταν τα τέσσερα λεπτά τα με, μεγαλύτερη διάρκεια όλης της προεδρίας μου. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ώρα τη νύχτα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Περνάμε στου αγορητέ που έχουν εγγραφεί. Είναι εκτενή ο κατάλογο των αγορητών. Πρώτο θα λάβει τον λόγο για ένα λεπτό. Πρώτη η κυρία η κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι εφόσον συζητούμε μια τόσο σημαντική έκθεση, νομίζω ότι οφείλω να ευχαριστήσω τον να θυμίσω εδώ στον εισηγητή ότι στο Δουβλίνο, ε, μπροστά στην αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή Ιρλανδοί Γεωργοί και σκοπεύουν να περάσουν εκεί τη νύχτα. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και δείχνει το πόσο απογοητευμένοι αισθάνονται τα μέλη τη γεωργική κοινότητα, οι ίδιοι Γεωργοί και οι καταναλωτέ, για την ασυνέπεια μεταξύ τη ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική και τη πολιτική τη για τα τρόφιμα και τη εμπορική τη πολιτική. Αυτό τονίζεται στην έκθεση αυτή. Είναι πολύ δυνατά τα επιχειρήματα που αναφέρονται εδώ. Κάποια φαίνονται να είναι ιδιαίτερα ε, απόλυτα, αλλά πραγματικά αντικατοπτρίζονται αναγνωρίζει την απογοήτευση που υπάρχει και από την απόψη των Ιρλανδών γεωργών. Πραγματικά πρέπει να δούμε ε, ε, εάν θέλουμε να κάνουμε τον τομέα αυτό ένα τομέα χαμηλών εισοδημάτων. Θα καταστραφεί το περιβάλλον μα έτσι. Να είμαστε συνεπεί και ω προ τι πολιτικέ τη ε, κλιματική αλλαγή. Το αποτύπωμα άνθρακα τη Βραζιλία, που βόει ο κρέατο τη Βραζιλία, είναι τετραπλάσιο από αυτού τη Ιρλανδία. διακόπτη πρόεδρο. Έληξε ο χρόνο σα. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριο Πυρίλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων ε, του πόρου αυτού που είναι πολύτιμο για τα κρατημέλη τη γεωργία και τη εμπορική πολιτική μα σε διεθνέ επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ χρειάζεται μια στρατηγική εμπορική η οποία να βασίζεται στι τάσει και τι δυναμικέ ε, τη παγκόσμια αγορά, αλλά και ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στον γεωργικό τομέα τη Ευρώπη. Αυτό ε, δίνει πολλά ωφέλη, όχι μόνο πολλά στην οικονομία, αντιμετωπίζοντα και το πρόβλημα τη ανεργία, αλλά ε, αν δεν λάβουμε μέτρα θα να έχουμε δυσκολίε ανάπτυξη σε κάθε περιοχή τη υπαίθρου μα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη γεωργική παραγωγή και να ευνοήσουμε τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τρίτε χώρε ώστε να έχουν τα ίδια πρότυπα ποιότητα ω προ την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την ευζοία των ζώων, των ανθρώπων και του κοινωνικού δικαίου. Σα ευχαριστούμε κύριε Πυρίλο. Τώρα ο κύριο Φεραίρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση που συζητούμε έχει πολλά παραδείγματα που αναφέρει για τις ολέθριε επιπτώσεις της απελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορίου στη Γεωργία. Η Γεωργία χρησιμοποιήθηκε ως ε, συναλλακτικό αντικείμενο για τις, ε, ε, τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου όμως δεν συνάγονται οι αναγκαίες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, στο παγκόσμιο εμπόριο που πρέπει να υπάρχει η λογική της συμπληρωματικότητας και όχι η λογική ανταγωνιστικότητας μεταξύ χωρών παραγωγών και χωρών καταναλωτών. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο προσανατολισμό όσον αφορά τι επιστημικέ ανάγκε κάθε χώρα. Μια γεωργία που θα βρίσκεται αντίθετη με την αναρχία της, των αγορών. Και πέρα από ε, ευλαβείς ε, δηλώσεις ε, και διακηρύξεις, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό είναι εκείνο το οποίο δεν ανέφερε η έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Η κυρία Νταϊάννα Ντότς τώρα παρακαλώ. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπω πολλοί από του συναδέλφου εδώ και ευχαριστώ τον συγκεκριτή για την έκθεσή του. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στι συνομιλίε μα στο τομέα του διεθνού εμπορίου. Εδώ, στη δική μα την εκλογική περιφέρεια, μπορεί να καταστρέψουν την κτηνοτροφία μα. Εδώ, στη Βόρεια Ιρλανδία, ακόμα και η βιομηχανία επεξεργασία μα απειλείται και εδώ. Το 16% του ΑΕΠ της περιοχής ε, ε, το καλύπτει η Γεωργία με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η ύφεση έχει προχωρήσει ε, ακόμη και στις ε, δυσχερέστερες οικονομικές συνθήκες. το μόνο που μας στηρίζει είναι ακριβώς η Γεωργία. Μπορεί να είναι ο κραγωνίος λίθος της οικονομίας μας και της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Η απελευθέρωση του εμπορίου και ιδίω οι τελευταίε συνομιλίε θέτουν σε κίνδυνο τι δεκάδε χιλιάδε αυτέ τι θέσει εργασία και την επιβίωση πολλών από του εκλογεί μα. Ευχαριστούμε κυρία Ντότ. Και τώρα ο κύριο Σον Κέλλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω πολλοί από τους Ολλανδού συναδέλφου και εγώ ανησυχώ ότι ο γεωργικό τομέα θα θυσιαστεί προκειμένου να ωφεληθούν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό είναι κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει. Πολλές από τις προτάσεις που γίνονται από την πλευρά τη Μαρκοσούρη είναι απαράδεκτες. Εδώ, χωρί να υπάρχει απαραίτητη διαβούλευση του Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να παίρνονται αποφάσει που καταστρέφουν την αγροτική βιομηχανία δεν θα υπάρξει αρκετή αντιστάθμιση ποτέ. Δεν μπορούμε να αντισταθμίσουμε μια κοινωνία για την απώλεια βασικών πόρων μια βιομηχανία που όλου του επηρεάζει στην κοινωνία, ιδίω στι γεωργικέ κοινότητε. Εδώ λοιπόν ανησυχούμε πάρα πολύ. Ε, όλο το θέμα των προτύπων της παραγωγής της Ευρώπης είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε καθημερινή, σε καθημερινή βάση η βασική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύσει το δικό της τον γεωλικό τομέα, εδώ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Ο κύριος Ταραμπέλα παρακαλώ. Θέλω να συγχαρώ τον συναδελφό Παστάμκο για την ποιότητα τη έκθεση, την οποία υπενθυμίζει τα βασικά κριτήρια που πρέπει να καθοδηγούν τον διαπραγματευτή τη Ένωση και τονίζει κυρίω τα μη εμπορικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται περισσότερο σε κάθε διαπραγμάτευση. Επίση, δεν είναι δυνατόν οι γεωργοί μα να αναγκάζονται να εφαρμόσουν τόσο αυστηρά πρότυπα για το περιβάλλον, εν υγιεινή, τη παραγωγή και αυτά όλα να θυσιάζονται στον φωμό του διεθνούς εμπορίου με τις τρευλώσεις του πάνω μπροστά στις τρίτες χώρες που μπαίνουν στην αγορά μας με προϊόντα που δεν σέβονται ακριβώς αυτόν τον τρόπο παραγωγής. Επίσης θα ζητούσα από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να επιδείξουν μεγάλη προσοχή στις συμφωνίες του Μερκοσούρ όχι μόνο ως την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία αλλά και ολόκληρη την ευρωπαϊκή γεωργία όπως το υπενθύμισε και ο εισηγητής διότι δεν δίνεται και για αυτήν καμία αποσημείωση στην αγορά. Ευχαριστούμε κύριε Ταραβέλα. Ο κύριος Σικέρσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Η εμπορική απελευθέρωση συνολικά έχει ωφέλη για διαφορετικούς εμπλεκόμενους και σε διαφορετικό βαθμό η γεωργική αγορά, η αγροτική αγορά είναι μια ειδική κατάσταση, διότι το κόστος παραγωγής εξαρτάται από το που παράγεται ένα προϊόν και αν η ποιότητα όσον αφορά τις απαιτήσει τηρούνται οι προδιαγραφές σε σχέση με τις απαιτήσει στην παραγωγική διεργασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υψηλότερες προδιαγραφές που καθιστούν τα προϊόντα που παράγουμε λιγότερο ανταγωνιστικά θα πρέπει να δούμε αυτές τις επιλογές ε, διότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τους καταναλωτές μας και την υγεία τους. Δεν θα πρέπει να είναι έκπληξη λοιπόν ότι ε, θα έπρεπε να αναμένουμε την ίδια αντιμετώπιση σε σχέση με προϊόντα τα οποία εισάγονται στις αγορές μας από τρίτες χώρες. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει υπερβολικά μεγάλες υπαναχωρήσεις ε, σε σχέση με τις ε, υποχρεώσεις που έχει αναλάβει εις βάρος των παραγωγών της. Ο κύριος Ταμπασδί παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να πω ότι αισθανόμαστε απογοήτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι όταν έρχεται η ώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερο εισαγωγέα τροφίμων παγκόσμια, αλλά και ο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκόσμια τροφίμων. Κάνουμε λόγο για ένα σύστημα παγκόσμιου εμπορίου που έχει απελευθερωθεί για παγκόσμιο ανταγωνισμό και είμαστε εμεί εκείνοι οι οποίοι επωφελούνται από αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με εκείνου του συναδέλφου που είπαν ότι έκανε κάποια πράγματα λάθο στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξετάζοντας το θέμα της εντολής και ο Διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν το είχε ομολογήσει έναντι μου σε σχέση με τι διαπραγματεύσει όσον αφορά προδιαγραφέ για το περιβάλλον, για τι απαιτήσει που είχαμε διατυπώσει. Δεν είχαμε το ίδιο επίπεδο απαιτήσεων έναντι των εταίρων μα. Υπήρχε κακή διατύπωση, υπήρχε κακή κίνηση σε σχέση με αυτά τα θέματα. Αναγνωρίζοντα ότι κάτι κάναμε λάθο στο παρελθόν, πρέπει να ξαναπροβληματιστούμε και να αλλάξει αυτή η εντολή. Γι' αυτό στο μέλλον πρέπει να διασφαλίσουμε οι εταίροι μα να κάνουν το ίδιο όπω και εμεί. Ευχαριστώ κύριε Ταμπαζή, λέει ο Πρόεδρο. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση τη κυρία Βέστλον, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το διεθνέ εμπόριο φυσικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ε, και οι συνομιλίε μα στον τομέα αυτό θα επηρεάσουν την δική μα γεωργική παραγωγή. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη και τι συμβαίνει ταυτόχρονα στην Αίγυπτο, στην Τινησία, στη Λιβύη. Οι εξελίξει στι χώρε αυτέ ε, έχουν απορροφήσει την προσοχή μα. Εδώ λοιπόν μια από τι σημαντικότερε ε, συνεισφορέ τη Ευρώπη θα ήταν να χρησιμοποιήσει τον τομέα που διαθέτει τόσο ισχυρό στην Ευρώπη, να, ε, να τον διαθέσει στου ανθρώπου αυτού που έχουν τόσα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ανησυχούμε για τι μεταναστευτικέ ροέ από τι χώρε αυτέ. Θα μπορούσαμε να φροντίσουμε οι άνθρωποι αυτοί να μην χρειάζεται να φύγουν από τι χώρε του, να μην ζητούν καταφύγιο σε εμά στο μέλλον. να του ενισχύουμε δηλαδή με τον γεωργικό μα τομέα εδώ μιλάμε για μια χώρα για τη χώρα μου, όπου έχουμε πολύ υψηλέ προδιαγραφέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υψηλότερε από οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι όπω το βλέπω εγώ, για τα πολιτικά και άλλα προϊόντα είναι χαμηλότερε. Σε ευχαριστούμε κυρία Βέσλοντ. Ολοκληρώνουμε έτσι αυτό το γύρο παρεμβάσεων. Με την τοποθέτηση τώρα στη συνέχεια τη κυρία Επιτρόπου, της κυρίας Δαμανάκη. Έχετε τον λόγο κυρία Δαμανάκη, παρακαλώ. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν δέχεται με χαρά την έκθεση αυτή. Ευχαριστεί τον εισηγητή κύριο Παπαστάμκο και τα μέλη και των δύο επιτροπών της Γεωργίας και του Εμπορίου για τις προσπάθειές τους να λύσουν συνοπτικά ένα πολύπλοκο θέμα. Μια σειρά συστάσεων της έκθεσης αυτής ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει και η ίδια η Κομισιόν που αναφέρονται σε πολλές μας ανακοινώσεις. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η απελευθέρωση του εμπορίου θέτει σημαντικές προκλήσεις για μας και για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά καθώς αναγνώρισε και το Κοινοβουλίο υπάρχουν και ευκαιρίες για τη Γεωργία από το διεθνές εμπόριο και τις διαπραγματεύσεις που το αφορούν. Επίσης πρέπει να δούμε ποια είναι τα ευρύτερα ωφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από το άνοιγμα του εμπορίου για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γενικά λοιπόν το σημαντικό θα ήταν να διατηρήσουμε το μήνυμά μας συνεπές. Το χρειαζόμαστε αυτό για να το εφαρμόζουμε σε όλες μας τις συμφωνίες είτε πρόκειται για την Τόχα με τους Αφρικανούς μας εταίρους είτε για το Μερκοσούρ. Γι' αυτό δεν θα ήταν σωστό να πούμε απλώς ότι το αυξημένο άνοιγμα του εμπορίου είναι απλώς ε, το χειρότερο ή το μικρότερο δυνατό σενάριο για την ευρωπαϊκή γεωργία. Οι εμπορικές συμφωνίες αντίθετα νομίζουμε δίνουν νέες ευκαιρίες από τις υποχωρήσεις των εταίρων μας. Και αυτό το στηρίζουν αριθμοί. Για το 2010 δείχνουν αυτοί ότι η Ένωση ως καθαρός εξαγωγέας αγροτροφημικών προϊόντων αντιπροσωπεύει πάνω από 90 δισεκατομμύρια και πάνω από 6 δισεκατομμύρια ωφέλει στο ισοζύγιό της. Αυτό εξηγείται από το στρατηγικό τονισμό που κάναμε στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων για τα οποία υπάρχει μεγάλη παγκόσμια ζήτηση και χάρη στην τεχνογνωσία του κάθε τροφιμικού μας τομέα συνεχίζουμε να παίζουμε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω, συμφωνώ και γι' αυτό Νομίζουμε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ τελευταία, τις τελευταίες δύο δεκαετίες βοήθησε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού, του γεωργικού τομέα ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς ενώ ταυτόχρονα η ποικιλότητα της γεωργίας στις χώρες της Ένωσης δεν παραγνωρίστηκε. Αν θέλουμε η Ένωση να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον των αγροτικών της περιοχών και με, μάλιστα με ισορροπημένο τρόπο και σε το περιβάλλον πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και επίσης ότι ιδιαίτερα ευαίσθητοι τομείς δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι θα διατηρήσουν υψηλό ρυθμό εισαγωγών χωρίς να πιεστούν ταυτόχρονα και οι τιμές. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όταν διαπραγματευόμαστε πολυμερείς συμφωνίες είναι επομένως να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της επιθετικής και της αμυντικής στρατηγικής μας καθώς και μεταξύ γεωργίας και άλλων υπολείπων τομέων του εμπορίου μας. Η Κομισιόν γνωρίζει πολύ καλά ότι έτσι είναι τα πράγματα και θα συνεχίσει σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο αυτά να φρονεί. Θα ήθελα λοιπόν να μας βοηθήσετε να κάνουμε, να πετύχουμε αυτή την ισορροπία για να δοθεί το σωστό μήνυμα και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Πίτροπε. Κλείνει εδώ, ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το σημείο. Θα ψηφίσουμε αύριο το μεσημέρι, 12.00 ώρα την αντίστοιχη πρόταση ψηφίσματος που μας ε, υποβάλλει ο εισηγητής κύριος ε, Παπαστάμκος και έτσι περνάμε στο ακόλουθο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι και το τελευταίο